Συνάδελφοι, κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Προπολογισμών και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Λάβατε τα πρακτικά των αποφάσεων των συντονιστών της συνεδρίασης της 23ης Απριλίου οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται στο φάκελο της συνεδρίασης και αν δεν έχετε αντίρρηση θεωρώ ότι τις αποδέχεστε. Αποδέχεστε τα πρακτικά. Και τώρα να καλωσορίσω εγκάρδια τον Επίτροπο Έτιγκερ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε που δεχτήκατε να έρθετε ήδη ε, σήμερα στην Επιτροπή των Προπολογισμών για να παρουσιάσετε με λεπτομέρειες αυτά που και χθες ε, ανακοινώσατε στην ε, Ολομέλεια και να σας πω πόσο το Κοινοβούλιο ε, παρατηρεί με προσοχή το γεγονός ότι εσείς ε, και εσείς και ο Πρόεδρος Γιούνκερ έχετε έρθει για να παρουσιάσετε τα στοιχεία αυτά ε, πρώτα στο Κοινοβούλιο και μετά στην παραδοσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι πραγματικά ένα δείγμα σεβασμού προς το Κοινοβούλιο που μας ε, συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη χθεσινή παρουσίαση του προπολογισμού και σας ευχαριστούμε και για τις διευκρινήσει που δώσατε κατά την παρουσίαση αυτή. Βεβαίω περιπλέκει κάπω τη συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ του πολιτου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και 2021-2027. Οπότε, Θα ακούσουμε με κάθε προσοχή και θα, θα δεχτούμε με κάθε προσοχή το σύνολο των εγγράφων που θα μπορέσετε να μας αποστείλετε ώστε να μην υπάρχουν αμφισημίες. Και όταν συγκρίνουμε ε, αριθμούς από το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το... σε σχέση με το καινούριο, να ξέρουμε ότι βασιζόμαστε ακριβώς στην ίδια βάση για να μην ε, χαθούν ε, κάποιες απορίες ή να μην εγερθούν κάποιες υποψίες. Και τώρα περνάμε σε μια φάση στενών διαβουλεύσεων, ελπίζοντας ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να ε, δώσει τη διαπραγματευτική του εντολή ώστε δυνατόν συντομότερα. Σε αυτή την ε, φάση, για την οποία αν υπομονούμε και θέλουμε να εργαστούμε, υπάρχει και ένας παράγοντας ε, εμπιστοσύνης και πίστης, για τον οποίο δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Γι' αυτό επιτρέψτε μου σύντομα και περιεκτικά να σας πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να αποσαφινιστούν πλήρως οι απορίες που ενδεχομένως να είχαμε ως τώρα για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μέσω της συνδιαλλαγής από το 2018. Ε, να μην υπάρξουν λοιπόν αμφιβολίες, θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό, ώστε να μην υπάρξουν σφάλματα. Ε, και παρανοήσεις. Από την δική μας την πλευρά δεν υπάρχουν αμφισημίες σε σχέση με όσα αποφασίστηκαν από εμάς και με τον έλεγχο του Γενικού Συγητή για τον Προπολογισμό του 2018. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να θίξω είναι η ε, διευκόλυνση ε, για την Τουρκία που αφορά του ε, Σύρου πρόσφυγε. Εδώ έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχε κάπω την εντύπωση ότι παραγωνίστηκε. Κάτι που δεν ε, συνηθίζεται και δεν ε, συνάδει και με τι διεκδικήσει μα. Να έχουμε ισότιμη μεταχείριση διότι η αρχή του προπολογισμού είναι διτή. το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Άρα θα δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε μια συμφωνία που δεν συνάδει ε, με την έγκριση τη δική μας στη δεύτερη δόση της διευκόλυνσης και εφόσον ε, για να δοθεί και η έγκριση του Συμβουλίου υπήρξε διορθωτικό του προπολογισμού με τη συνήθεια διαδικασία και πέρασε και από τις σκληρές διαπραγματεύσεις που συνήθως οργανώνται μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Με αυτά λοιπόν θα ήθελα να επιμείνω, Επίτροπε, στην ε, πρόθεσή μας να εργαστούμε σκληρά μαζί σας ε, και με την ομάδα των συνεργατών σας σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και χωρίς ε, επιφυλάξεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που θα μας παρουσιάσετε τώρα όσα δεν μπορέσετε να μας πείτε χθε στην Σύνοδο Λομέλειας. Μπορούμε τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ο καθένας γνωρίζει ότι συχνά ο διάβολος ακριβώς εκεί κρύβεται, στις λεπτομέρειες. Αλλά ας κοιτάξουμε μαζί να τον βγάλουμε εκτός παιχνιδιού, ώστε να είναι ε, καρποφόρες οι διαπραγματεύσει μας και όπως ξέρουμε και το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε αυτά που ενέκρινε, οπότε το Κοινοβούλιο από την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων και για το πλαίσιο του 2021-2027 πρέπει να κοιτάξει να καλύπτει τις προσδοκίες και των κυβερνήσεων των 27 μεν αλλά και των ίδιων των πολιτών, των Ευρωπαίων που εμείς ως βουλευτές εκπροσωπούμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε την ευκαιρία τόσο γρήγορα μετά την παρουσίαση της πρότασης μας για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις πρώτες συζητήσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε μαζί και μπαίνουμε έτσι στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η πρώτη φάση ήταν η φάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλουτίσατε την πρόταση με πολλές επαφές και συναντήσεις εδώ ε, με την Επιτροπή σας, άλλες επιτροπές, με τον Πρόεδρό σας, το Προεδρείο και δύο εκθέσεις τις οποίες μελετήσαμε και φροντίσαμε και προσπαθήσαμε ε, να τις συμπεριλάβουμε στις προτάσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Σήμερα το πρωί, δύο μισή ώρες, ε, συζητήσαμε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, στην ΚΟΡΕΠΕΡ, με τους πρέσβες στο Συμβουλίο, και τους δικούς μας και τους δικούς σας πρέσβεις, τους οποίους γνωρίζετε όλοι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωινή συνεδρίαση. Είναι σαφές ότι εδώ στο Κοινοβούλιο αγωνίζεστε για κάθε ψήφο, αλλά εκεί αρκεί μια πλειοψηφία. Και εμεί αγωνιζόμαστε στο Κορεπέρα, αλλά και χρειαζόμαστε όλες τις ψήφους. Από την Κορεπέρα μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εχθές πολλά κράτη και πολλές κυβερνήσεις έκαναν σχόλια, tweets, τα διάβασα όλα. Τα πρώτα έφτασαν ήδη πριν καν αρχίσει τις συζητήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι λαθασμένη κίνηση, ξέρετε. Η πρώτη επιτρέπεται, στη δεύτερη αποκλείεσαι. Το θέμα είναι πώς θα συμφωνήσουμε. Η πρότασή μου δεν είναι το απάβγασμα της τελειότητας, ούτε το τέλος μιας συζήτησης. Είμαι υπέρ ε, της συζήτησης να μου πείτε καλύτερα επιχειρήματα, ε, πού θα κάνουμε περικοπές, οικονομίες, ε, ανακατατάξεις κτλ. Εγώ δεν είμαι μέτοχος του προϋπολογισμού, εγώ είμαι ο διαμεσολαβητής, ο συντονιστής. Εσείς είστε στη θέση του οδηγού και το Συμβούλιο. Γι' αυτό συνιστώ να έχουμε προσέγγιση ευέλικτη και να κοιτάξουμε τι θα γίνει με την έρευνα, την ε, διευκόλυνση ε, συνδέοντας την Ευρώπη, τη συνοχή, τα γεωργικά. Ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε όλο το πακέτο. Αν ο καθένας προτείνει τα δικά του συμφέροντα και ενδιαφέροντα με άκαμπτο τρόπο, δεν γίνεται δουλειά. Το αντίθετο, εάν υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας και ευελιξίας, θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι περίπλοκος ο στόχος μας. Κάναμε μια πρόταση για άλλη μια επταετία και εξαγγείλαμε ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μεθεπόμενη θα οφείλει να κάνει πρόταση για μια πενταετία ή πέντε συν πέντε έτη. Είναι σαφή τα ε, επιχειρήματα. Αυξήσαμε και τους τίτλους. Μέχρι τώρα ο μέσος πολίτης δεν μπορούσε να κατανοήσει ε, τι είναι αυτοί οι πέντε τίτλοι ή ο τίτλος ένα α και ένα β κτλ με τους τίτλους τώρα ε, έχουμε δημιουργήσει ε, ορατότητα για την πολιτική και έχουμε νέους τίτλους για ε, κάποιες αρμοδιότητες που μέχρι τώρα δεν ήταν ευρωπαϊκές ή περιορισμένα μόνο. Η ασφάλεια και η άμυνα, μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων. Και επειδή πολλοί πολίτες και πολλά κράτη-μέλη μας έλεγαν ανέκαθαν ότι έχουμε υπερβολικά πολλά προγράμματα. Μια ζούγκλα ε, ολόκληρη. Και ανά πενταετία συνεχίζαμε ε, τα προγράμματα που υπήρχαν και προσθέταμε και καινούρια ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν ή του Συμβουλίου. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να συνενώσουμε κάποια προγράμματα για να αυξηθεί και η ευελιξία και να κάνουμε έτσι κλάστερς και να απλοποιήσουμε τους κανόνες που τα διέπουν. Όλα αυτά, λοιπόν, οι τίτλοι έχουν γίνει 7 πλέον, όχι 5, 38 τα προγράμματα και όχι 57, ε, ενωμένα προγράμματα. Αυτό τώρα καθιστά δυσκολότερη τη συγκρισιμότητα. Εντάξει, όταν έχεις 100 προγράμματα και δεν αλλάζεις τίποτα, ε, μπορείς να τα συγκρίνεις, γιατί συγκρίνεις τις γραμμές του προπολογισμού στα τευτέρια. Αλλά αυτό δεν είναι σωστή πολιτική. Θα πρέπει να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Έχουμε νέε ευθύνε για τη μετανάστευση, για την αναπτυξιακή βοήθεια, για τη φύλαξη και διαχείριση των συνόρων, για την αμυντική έρευνα. Θα πρέπει να υπάρχει χώρο στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί πρόκειται για το μέλλον τη Ευρώπη. Συγκρισιμότητα τι σημαίνει. Ότι έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Τα νέα προγράμματα είναι λιγότερα και νέα κέντρα βάρους. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι το βλέμμα προς το μέλλον στραμμένο. Εκεί έχουμε εστιάσει την προσοχή μας. Είμαι πεπισμένος ότι η έξοδος των Βρετανών θα έχει συνέπειες και πρέπει να έχει συνέπειες στον προπολογισμό. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε και να υποδιόμαστε ότι μπορούμε να ε, χρηματοδοτούμε όσα τα προγράμματα έχουμε και άλλα περισσότερα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα μείγμα ανάμεσα σε περικοπές και υψηλότερες εισφορές. Κάποια κράτη-μέλη παραμένουν στο 1,0% ότι θα θεωρούν οροφή του ΟΕΠ Και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούν δευτερεύοντα. Εμείς προτείναμε 1,114. Δεν ακολουθούμε πλήρως την πρόταση του Κοινοβουλίου, αλλά κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση του Κοινοβουλίου και πιστεύουμε ότι τα περισσότερα χιλιοστά ή περισσότερα ποσοστά θα οδηγήσουν σε ακόμα σφοδρότερες ή θα οδηγούσαν σε ακόμα σφοδρότερες αντιστάσεις και αντιρρήσεις στα κράτη-μέλη και θα δυσκόλευαν έτσι ε, περαιτέρω τις ε, πιθανότητες που θα είχαμε να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Αύριο θα δω ε, τη βαβαρική κυβέρνηση. Εγώ την αγαπώ τη Βρετανία. Αλλά 1,3% αν το ψηφίσει βαβαρός θα πρέπει να ζητήσει άσυλο στις Βρυξέλλες. Και την Αυστρία την αγαπάω. Αλλά ξέρετε, Εσείς έχετε διπλή ιδιότητα κάθε φορά. Είστε και ευρωβουλευτής, αλλά και του κράτους μέλους σας. Και του κόμματός σας, του δημοκρατικού που εκπροσωπείτε εδώ. Αυτό που ζητάτε εδώ συνδυάζεται με το περιθώριο λιγμό που έχετε στη χώρα σας. Δηλαδή στη Βιέννη να λέμε 1,3% 1% ε, και στις Βρυξέλλες 1,3%. Μα δεν γίνεται, χρειάζεται μια μέση οδός. Η οροφή δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στο σκοπό μας. Ένα μέσο για να φτάσουμε στο σκοπό μας. Για προγράμματα πρόκειται εδώ. Άρα, ας κοιτάξουμε όλα τα προγράμματα και μετά να ελέγξουμε. Η πρόταση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρκεί για να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι περικοπές είναι περιορισμένες, είναι μετριοπαθείς, είναι κάτι που μπορούμε να αποφασίσουμε. Και πού κάνουμε λάθος στις αποφάσεις για την ε, ανάπτυξη και για την έρευνα. Τα δύο μεγάλα προγράμματα παραμένουν, τα δύο μεγαλύτερα, η συνοχή και η κυνηγεωρική πολιτική. Ε, παραμένουν να καλύπτουν περίπου 30% του δημοσιονομικού μας πλαισίου. Οι περικοπές στη συνοχή είναι της τάξεως του 6,2%. Ε, ας πούμε 7. Ε, για τις γεωργικές λίγο κάτω του 5%. Οι άμεσες πληρωμές είναι λιγότερες κάτω του 4%. Και αυτό μπορώ να βγω να το πω σε οποιαδήποτε συνομοσπονδία γεωργών, σε οποιοδήποτε αγρότη και όποιο μου ε, στο κοινοβούλιο. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν και οι αγρότες ότι το Brexit αλλάζει τα δεδομένα. Είμαστε με μείον 4%, μείον 5%, μείον 6% και παρόλα αυτά είμαστε στο πλευρό των περιφερειών της υπαίθρου και του αγρότη. Και για τα δύο προγράμματα δεν έχουμε κάνει τη συνολική πρόταση. Σας παρακαλώ δώστε μας χρόνο μέχρι τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου για να ε, σας υποβάλουμε τις εκτελεστικές ε, διατάξεις για τη συνοχή και για τους δύο πυλώνες της Γεωργίας, για να δούμε συγκεκριμένα ποιες επιπτώσεις θα έχουν τα νέα μας δημοσιονομικά σχέδια για την Ήπεθρο, για τον Αγρότη, για την Περιφέρεια και για την κοινωνική πολιτική. Θα ξανάρθω με τους συναδέλφους Κρέτσου και Χόγκαν για να υποβληθώ στη ε, δική σας ε, κρίση. Θέλαμε με την πρόταση αυτή του προπολογισμού να στραφούμε προς το μέλλον της Ευρώπης και να δείξουμε κάτι που το 2011 δεν ήταν ακόμα ευρωπαϊκή υπόθεση ούτε ευρωπαϊκό ε, πρόβλημα η μετανάστευση το 2011 δεν ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε σε αυτό ε, το μέγεθος. Δεν είχαμε φίλιο στη Συρία, δεν είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή. Η Αραβική Άνοιξη ήταν ελπίδα και όχι χήμερα ακόμα. Η γειτονία μας ήταν πολύ πιο σταθερή και γι' αυτό στη γειτονία πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στους ανθρώπους, στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, ενώ στο εσωτερικό της Ευρώπης ε, με τη μετανάστευση και την εσωμάτωση πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Και, και τα κράτη-μέλη που θίγονται περισσότερο, που δεν είναι η Ιρλανδία, δεν είναι μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Βουλγαρία. Να τους δώσουμε, να τους λοιπόν διοικητική βοήθεια και οικονομική βοήθεια. Και ακόμα. Αυτό ακριβώς ε, τώρα που υπενθυμίσε ο κ. Ε, Μπέγκε ήταν και ένα θέμα που πρότεινε η Κομισιόν στην ε, τελευταία πρόταση του προπολογισμού και του Κοινοβουλίου άλλωστε, αλλά απλά το απέρριψε το Συμβούλιο τότε. Και το ίδιο ισχύει και για το Connecting Europe, για την ψηφιακή υποδομή, τότε η Νέλη Κρούς είχε προτείνει 1,5 δισεκατομμύρια. Τι έκανε το Συμβούλιο, 1 δισεκατομμύριο. Σήμερα γνωρίζουμε πως ήταν μεγάλο λάθος. Και πάλι ανέβηκε το ποσό στα 9 δισεκατομμύρια. Δικαίως, γιατί θέμε τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και υπολογιστέ υψηλών επιδοσών και πραγματικά αναμένω την αντίδραση αυτή τη φορά. Και μετά μιλάμε για Silicon Valley, Huawei, Alibaba και δεν μπορεί η Ευρώπη να ακολουθήσει. Το μέλλον λοιπόν σημαίνει καινοτομία, σημαίνει έρευνα, σημαίνει ανάπτυξη. Σημαίνει 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία. Αυξάνουμε λοιπόν τον ορίζοντα κατά πάνω από 60%. Πάνω από 60%. Αν λοιπόν περικοπούν αυτά, υπονομεύεται το κοινό μας μέλλον. Με το να συνδέσουμε λοιπόν αυτά τα κονδύλια με τα κονδύλια της συνοχής δίνουμε την δυνατότητα στα κρατη που δεν έχουν τόσο μεγάλες ερευνητικές δυνατότητες την δυνατότητα να μετατοπίσουν κονδύλια από την συνοχή στην έρευνα και έτσι να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τις περιοχές που είναι πιο ισχυρές στην έρευνα όπως το Παρίσι, η Λιόν, η Ιρλανδία, η Βαβαρία, η Βάδη, Βιρτεμβέργη κτλ. Έχουμε διπλασιάσει το Εράσμος. Θεωρώ πως μια απάντηση στον ευρωσκεπτικισμό μπορεί να είναι οι νέοι της Ευρώπης κατά τη διάρκεια τη εκπαιδευσής τους των σπουδών του να έρχονται σε επαφή με άλλου πολιτισμές, άλλες γλώσσες, άλλη φύση, άλλη αγορά εργασία, άλλη μουσική. Θεωρώ ότι έτσι ή ε, ο διπλασιασμός είναι μία απάντηση. Κάποιοι μίλησαν και για τριπλασιασμό. Συν 60% λοιπόν στην καινοτομία, συν 100% στο Εράσμους και αύξηση των κονδυλίων για την γειτονία και τον κόσμο για την αναπτυξιακή βοήθεια, αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό και μετά. Όμως θα πρέπει να δούμε το θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων μαζί με τα πληττόμενα κράτη. Και αυτό για να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε έναν χώρο Σέγγεν χωρίς εσωτερικούς ελέγχους. Οπότε η Frontex από 1.200 άτομα θα πάει στα 10.000 άτομα. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι business as usual. Μιλάμε για πλήρη ανατροπή και εξυγχρονισμό του προϋπολογισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αποστολές της Ευρώπης της επόμενης δεκαετίας. Το Κοινοβούλιο ήταν και είναι και θεωρούσε βεβαίως σημαντικό να αλλάξει και η πλευρά των εσόδων. Και αυτό κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ένα διψήφιο, υψηλό διψήφιο νούμερο δισεκατομμυρίων στην πλευρά των εσόδων από τους ίδιους πόρους. Κάτι το οποίο θεωρώ και σημαντικό ψυχολογικά γιατί όταν είναι οι εθνικοί βουλευτέ υπεύθυνοι για το 70% των εσόδων μας και χρειάζεται να του παρακαλάμε, αυτό δημιουργεί μια αίσθηση I want my money back που λέγει η Θάτσερ, μια λάθος νοοτροπία. Γι' αυτό έχουμε και το δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας για τα έργα της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας τα πλαστικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αφετηρία για μια εισφορά των κρατών μελών και να υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για εισφορές μέσω εθνικών φόρων στα προϊόντα συσκευασίες και στα πλαστικά εκείνα τα οποία δεν ανακυκλώνονται. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μπορείτε να διαβάσετε ούτως ή άλλως την ε, πρόταση μονη σας. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ερωτήσεις σας και η κριτική σας. Και είμαι σίγουρος ότι θα πηγαίνει προς την τελείως αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την οποία άκουσα σήμερα το πρωί. Βεβαίως, αν δέχομαι πειρά από παντού, τότε σημαίνει ότι κάνω σωστά την δουλειά μου. Από αριστερά, δεξιά, από συμβούλιο, κοινοβούλιο, αν υπάρχει σωστή αλλά δίκαιη κριτική, σημαίνει ότι σωστά κάνω. Αυτό το οποίο πρέπει. Κάτι τελευταίο. Σήμερα στον τύπο υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια που ήταν ουσιαστικά και πολλές τοποθετήσεις κρατών μελών που εστίασαν στην αύξηση των συνεισφορών. Παραδείγματος χάρη, στην ε, χώρα μου μιλάνε για μια αύξηση από 11 έως 12 δισεκατομμύρια. Σε τι ε, βασίζονται. μιλάμε για έναν προπολογισμό του 2019, σε σύγκριση με το 2018 έχει μια αύξηση 2-3%. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Το πρόβλημά μα λοιπόν είναι ότι εμεί καταρτίζουμε μακροπρόθεσμο προπολογισμό. Γιατί οι ερευνητέ, οι περιφέρειες, οι γεωργοί, οι δήμαρχοι θέλουν να χρηματοδοτήσουν έργα που θα υλοποιηθούν σε 5, 6, 7 χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια σχεδιασμού. Αλλά αν συγκρίνουμε το 2014 με το 2027 είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Σε αυτά τα 14 χρόνια έχει έχουν αυξηθεί οι μισθοί των ερευνητών, η τιμή της βενζίνης, οι τιμές ε, για τα έργα, τα δομικά, για τα έργα τα στερεοδρομικά. Έχουν διπλασιαστεί. Δηλαδή είναι σαν να συγκρίνουμε έναν προπολογισμό της εποχής του Χάλσταϊν, της Κομισιόν του Χάλσταϊν, με τον τωρινό βεβαίως, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Και αν συγκρίνουμε σε 20 χρόνια στο μέλλον, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Γι' αυτό η παράκλησή μου είναι εξή. Να μεταφέρετε το εξή μήνυμα. 7 χρόνια. Επί τον ετήσιο προπολογισμό 1,6-1,7. Είναι 12-13% ονομαστική αύξηση. Χωρίς να σημαίνει κάτι το περισσότερο. 7 χρόνια ανάπτυξη του ΑΕΠ 1,82%. Είναι συν 17%. Οπότε αυτομάτως ονομαστικά μιλάμε για 30% παραπάνω εισφορές χωρίς να μιλάμε για κάποιο περισσότερο προϊόν τελικά. Δηλαδή αυτή την αύξηση τη χρειαζόμαστε για να παραμείνουμε στο ίδιο σημείο εσόδων και εξόδων. Με αυτά τα δύο μόνο δηλαδή, αύξηση του πληθωρισμού και του ΑΕΠ για αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα ίδια ισχύουν βεβαίως και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα δούμε. Τις επόμενες ημέρες θα βρω τα στοιχεία των προϋπολογισμών μέχρι το 2027 όλων των κρατών μελών, ειδικά για αυτά τα οποία ασκούν ιδιαίτερη κριτική. Και εκεί πέρα θα δείτε ότι μιλάμε για αυξήσει 30-40%. Γιατί ε, παραμένουμε στο ένα ακόμα κάτι του ΑΕΠ. Και αυτομάτως υπάρχει αυτή η ονομαστική αύξηση, αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Το Brexit και τα 11 ή 14 εκατομμύρια τα οποία δεν θα τα βρούμε μόνο από περικοπές. Ή έχουμε τις ε, νέε αποστολές, τη μετανάστευση, την προστασία των συνόρων. Δεν μπορούμε τους ανθρώπους που θα πάνε στα σύνορα να τους πληρώσουμε με καλά λόγια. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί κοστίζουν 60.000 ανά άτομο, ανά έτος. Επί 10.000 άτομα αντιλαμβάνεστε το ποσό. Οπότε μιλάμε για μια αύξηση η οποία είναι πραγματική εν μέρη και εν μέρη ονομαστική. Και έχουμε από τη μία μια χώρα σαν την Γερμανία η οποία πληρώνει αυτή τη στιγμή 25 δισεκατομμύρια το έτος και θα αυξηθεί αυτό σε 36 δισεκατομμύρια το έτος στο επόμενο πηδελταπή. 7 όμως από αυτά τα δισεκατομμύρια από την αύξηση των 11, είναι, των 11 δισεκατομμυρίων είναι αύξηση λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ. Οπότε σας παρακαλώ ασκήστε μου κριτική, λεπτομερή αλλά να δείτε τα στοιχεία και να μην απορρίψετε τον προϋπολογισμό στον ε, σύνολό του, την πρόταση αυτή. Και ελάτε σε επαφή με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Ευχαριστώ. Merci, merci, monsieur le commissaire. Ευχαριστώ κύριε ε, Αν θέλετε θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον εισηγητή μα, στους συνεισηγητές για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά τους συνεισηγητές για τους νέους ιδίους πόρους. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε στις 3.30, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε ανελημμένες υποχρεώσεις, παρακαλώ να σεβαστείτε όλο το χρόνο αγόρευσή σας που θα είναι δίλεπτος. Ο Γιάννη Ολμπριχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πώς κάνουμε συμβολικά και παραδοσιακά, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχουμε μια νέα αρχή. Ε, αρχίζει μια νέα φιλοσοφία να εφαρμόζεται στον προπολογισμό. Το βρίσκω αισιόδοξο λοιπόν αυτό και συνεχίσουμε να το σκεφτόμαστε έτσι. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε ταυτόχρονα είναι μεταξύ του 1,0 και 1,3 να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας μια ξεκάθαρη θέση. Αλλά ε, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και πρέπει να το πω σε εισηγητής της Επιτροπής Προπολογισμών είναι μια σαφής εξήγηση για τους αριθμούς. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να καταλάβουμε τι εννοείται με την πρότασή σας. Εννοείται όταν λέτε 1,3 από τη δική σας πλευρά ε, τι πρέπει να κάνουμε, τι θα κοστίσει και ποιο θα είναι το επίπεδο, αυτό αναλύεται. Διότι περιμένουμε κάποια αντίδραση, ε, μια απάντηση να μας λέει ξεκάθαρα τι έχει υπολογίσει τι θα κοστίσει και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Διότι δεν είναι η συζήτηση μόνο το 1,3 και φτάνει. Ε, μπορεί να θέλετε να γίνει μια μείωση, εντάξει, αλλά πού θα γίνουν οι περικοπές, από ποιες δράσεις είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χρησιμοποίησατε πολύ στρογγυλεμένους αριθμούς, όπως 5,5, 5,6, ακόμη και για τη συνοχή χθε είπατε κάτι για 7. Άρα Θέλουμε να δούμε τη συλλογιστική σας. Δεν είναι το πρόβλημα το 1,1-1,3. Είναι θέμα τι θα κοστίσει ακριβώς και τι θέλετε να κάνουμε συγκεκριμένα. Έτσι εργαζόμαστε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Θέλουμε ακριβείς αριθμούς. Πάντως ε, για τις ε, πρώτες αντιδράσεις μας να πω, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε με απλό τρόπο. Μείον 5 ή μείον 6 για την συνοχή και τη γεωργία. Για ποιε αξίες μιλάμε Ποιο είναι το 100%? Υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις. Άλλοι μετράμε τους πληθωρισμούς και λέμε δεν είναι 5, είναι 15. Άλλοι λέμε δεν είναι 15, είναι 10. Το μείον 5, μείον 6 σε τι ακριβώς αναφέρεται. Και επίσης το άλλο που πρέπει να πω είναι για την ερεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Ναι. Αλλά ως εισηγητής, συνεισηγητής, πρέπει να πω ότι αυτό που χρειαζόμαστε από εδώ και μπρο είναι ε, συγκεκριμένοι αριθμοί και τι ακριβώς σημαίνουν. Τι εννοείται και τι ακριβώς θα κοστίσει. Ευχαριστούμε κυρία Τομά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Όπως σας είπα και χθε, απογοητεύτηκα ιδιαίτερα από την πρότασή σας, αλλά σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Και θα ήθελα να συμμεριστώ την αισιοδοξία του συνεισηγητή μου. Και ελπίζω αυτή η αισιοδοξία να πλωθεί σε όλη την Επιτροπή Προπολογισμού, γιατί η μάχη μόλις ξεκινάει. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. Όμως για να ξεκινήσει πραγματικά η μάχη. Θα πρέπει εμεί στην Επιτροπή Προπολογισμών να καταλάβουμε. Και όπω είπε ο συνάδελφο, έχουμε πρόβλημα με του αριθμού. Συγκεκριμένα. Για να σας εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πολύ απλά αριθμούς για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 στις τιμές του 2018. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση εάν πάρουμε τον προπολογισμό τον επόμενο με τις τιμές τις σημερινές και δεν κάνουμε αυτή την αντιπαραβολή. Θα πρέπει αυτό να είναι το πύχη βάσει την οποία θα κάνουμε όλες τις υπόλοιπες συγκρίσεις. Και έχουμε και ένα μικρό πρόβλημα πληθωρισμού. Νομίζω ότι τον εκτιμήσατε σε υψηλότερα επίπεδα για τα ερχόμενα χρόνια και αυτό ήταν και κάτι σαν τέχνασμα που το ανέφεραν και κάποιοι αυστριακοί εκπροσώποι σε κάποιες από τις συνεδριάσεις. Όσο πιο υψηλά τα υπολογίσουμε, τόσο πιο διαφορετικά μπορούμε να υπολογίσουμε και τα ποσά που παρουσιάζονται. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις του πληθωρισμού γιατί δεν είναι βέβαιες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορούμε να εργαζόμαστε σοβαρά, διότι αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία και μας λείπουν προς στιγμήν. Λείπουν για να μπορέσουμε να κάνουμε μία ακριβή ανάλυση, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την παρουσίαση σας και όσο μας είπατε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Και να σας πω, Επίτροπε, ότι εδώ δεν είμαστε χωρισμένοι σε βορρά και σε νότο. Εδώ είμαστε Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει πλειοψηφία 458 βουλευτών που ψήφισαν το ίδιο σχέδιο προπολογισμού για το 2021 ως 2027. Δεν ε, σκεπτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Άλλο το Συμβούλιο και άλλο το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είμαι ιδιαίτερη αισιόδοξη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα ως συνσηγητής για τους νέους ιδίους πόρους. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Αυτό το συζητάμε πιο εύκολα με γραπτά α, μπροστά μας, αλλά όπως είπαν και οι δύο συνεισηγητές, ο τρόπος αυτός της ε, Κομισιόν για την ε, παρουσίαση είναι αρκετά έξυπνος, αλλά όχι αρκετά διαφανής για όσους θέλουν να συγκρίνουν, γιατί θα έπρεπε να μιλάμε για τιμές 2018 και το ίδιο και για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Το καλό είναι ότι έχουμε άλλη μία προσπάθεια για να απλοποιήσουμε την πλευρά των εσόδων. Ο ΦΠΑ τώρα είναι απλούστερος χωρίς τους Βρετανούς. Φορολογία επιχειρήσεων μας δίνει ε, το μισό από αυτό το ποσό. Για το ETS, το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών ε, για κάποιες χώρες είναι εκτός συζήτησης ε, και θα συνεισέφερε ούτως ή άλλως το 2% των μελλοντικών εσόδων. Επίσης κάποιοι υποψήφοι είναι ψηφιακός φόρος και φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Καλό το ότι μας υπόσχεστε και άλλα ε, και άλλες πηγές ε, εσόδων και να αφαιρεθούν οι διορθώσεις και οι επιστροφές όμως δεν σημαίνει ότι κάθε διορθώση σχετίζεται με την Βρετανική επιστροφή, να δούμε αν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε μια τρίτη θέση για τους καθαρούς εισφορείς χωρίς κάποιες διορθώσεις. Ε, είμαι επιφυλακτικός ως προς αυτό, γιατί βεβαίως οι συνάδελφοι ε, ε, ξεχνάνε ότι έχουμε και πάρα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Το κόστος μείωσης δεν είναι το καλύτερο μήνυμα για τον συνεισηγητή μου έπεσε από το 25% στο 20%. Λοιπόν, στο Κοινοβούλιο είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι για δράση για να μεταρρυθμίσουμε την πλευρά των εσόδων. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Επί του παρόντος, πέντε αιτίες για ικανοποίηση, μια ανησυχία και μια δυσφορία δυσφορία. Υπάρχει, μάλλον η πρώτη ικανοποίηση, έχουμε ιδίου πόρου, πολύ ωραία, δεν υπήρχε στο παρελθόν δεύτερο, προτείνεται μια δέσμη και ανέκαθεν εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι δέσμη για να υπάρχουν κάποια αντισταθμίσματα ε, από κατηγορία σε κατηγορία. Τρίτον, νέοι ήδη πόροι και στην έκθεση Μόντι το έλεγε αυτό και στη δική μας έκθεση του κυρίου Λεβαντόφσκη και μου και το υιοθετήσατε. Μπράβο σας. Τέσσερα. Οι νέοι ήδη πόροι ανταποκρίνονται σε δύο στρατηγικούς στόχους που όλοι εκτιμούμε. Είναι η βελτίωση σωστή της εσωτερικής αγοράς ο ένας και ο δεύτερος προστασία του περιβάλλοντος και καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Και τέλος, το είπε τώρα μόλις και ο Γιάννους Λεβαντόφσκι, προτείνεται να καταργηθούν οι επιστροφές, αν και το χρονοδιάγραμμα για ορισμένα πράγματα ε, εντάξει, ξέρουμε. Ποιο είναι, ποιος είναι ο ρυθμός που θέλετε να προχωρήσετε για τους ιδίους πόρους. Ανάλογα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν οι εθνικές εισφορές. Τώρα, γιατί είμαι δυσαρεστημένος. Το ποσό γενικά δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα θέλαμε και το κέντρο βάρους παραμένει, από ό,τι φαίνεται, στις εθνικές εισφορές. Δεν ναι, μας ικανοποιεί καθόλου αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους πόρους και τα έσοδα, δεν έχετε λύσει το πρόβλημα των προστήμων που πληρώνουν οι εταιρείε που θα μπορούσε να τροφοδοτεί τον προπολογισμό των δεφών κρατών μελών. Απλώς μας λέτε ποια είναι τα έσοδα από την υλοποίηση κάποιων πολιτικών με τα πρόστιμα τι γίνεται και για ποιο λόγο δεν το αναφέρετε. Ευχαριστώ. Sí. Ευχαριστώ και εγώ. Προχωρούμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής Προπολογισμών, ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Κάθε φορά που το συζητάμε, νομίζω ότι η σωστή πρόταση είναι αυτή του Κοινοβουλίου. Έχουμε μια πρόταση την οποία την προασπιζόμαστε. Δηλαδή, να υπάρξουν μειώσεις μόνο ε, στη συνοχή και στη γεωργία και με τις προτάσεις που έγιναν στο, με τις αυξήσεις μάλλον που έγιναν στο Erasmus Plus και στο κόσμο. Εδώ ε, το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει άλλε προτάσει. και αν ε, το Συμβούλιο δεν δεχτεί τις προτάσεις της Επιτροπής ε, θα περάσουν περικοπέ στη Γεωργία και τη συνοχή που θα είναι διαφορετικέ. Εδώ λοιπόν αυτό αποτελεί πηγή δυσαρέσκεια για μας. η ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα είναι κάτι που το θέλουμε, είναι θετικό. Όμω σημειώνω ότι υπάρχει μια σαφής ρήξη σε σχέση με την εσωτερική αλληλεγγύη τη Ένωση από την προοπτική του προπολογισμού. Οι περικοπέ πρέπει να γίνουν με πολύ προσεκτικό και συγκεκριμένο τρόπο. Και να κάνω εδώ μια ε, παρέκβαση. Ε, ξέρουμε ότι είναι το Κοινωνικό Ταμείο, το, το Ταμείο Συνοχή και το ΦΕΝΤΕΡ η πολιτική συνοχή. 5% ε, ήταν οι αριθμοί που αναφέρθηκαν. 6,2 εδώ, 5% ήταν στο, 5 ήταν στο αρχικό κείμενο, φτάνουμε το 10%. Ίσως τελικά τι περικοπή θα γίνει. Ελπίζω λοιπόν ότι η πολιτική της συνοχής δεν θα αποτελέσει παράδειγμα που θα ε, γίνει πηγή, ε, χαρτοφυλάκιο για να ε, χρηματοδοτήσουμε τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Όχι, κοινωνικό ταμείο, ταμείο συνοχής και φεντέρ. Αυτά είναι η βάση της πολιτικής συνοχής. Και εδώ χρειάζεται μια τεχνική συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου, διότι πρέπει να συνεννοηθούμε. Τα μαθηματικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι διαφορετικά. Μην μιλάμε για ε, διαφορετικά πράγματα ενώ λέμε τα ίδια. Και μια και μιλάμε για μείωση τη αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε σε αυτόν τον προπολογισμό σε σχέση λόγου χάρη με το Ταμείο για τη Σταθεροποίηση την ε, οικονομική σταθερότητα. Αυτό λέει θα μείνει εκτός προπολογισμού και θα υπάρχουν ε, κονδύλια που θα είναι ήδη ε, προκαθορισμένα για αυτό το στόχο και για να υπάρχει σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής πολιτικής και για την τομή της ανάπτυξης. Είμαστε υπέρ του να βρίσκεται μέσα στον προπολογισμό, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια αύξηση, μια ενίσχυση. Διότι αν πρόκειται να μπει μέσα, αλλά να γίνουν περικοπές σε άλλες πολιτικές, καλύτερα να το είχαμε κρατήσει έξω από τον προπολογισμό για να μην τον υπερφορτώσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν για τη μουσονομική πειθαρχία που προσπιζόμαστε αλλά θα πρέπει όλα αυτά να ανταποκρινόνται και στις σωστές αυξήσεις και ενισχύσεις. Και επίσης, μια τελευταία κουβέντα. Όλα τα κράτη-μέλη είναι δικαιούχοι του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, ε, γνωρίζουν μεγαλύτερες ανισότητες. Κάποια από αυτά ε, τα είδαμε πρόσφατα και με τα προγράμματα προσαρμογής. Ελπίζω λοιπόν ο προπολογισμό να συμβάλλει στην εδαφική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τις οποίες δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε καμία περίπτωση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που ήρθατε στην Επιτροπή μα για άλλη μια φορά να μας μιλήσετε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπαν πολλοί εισηγητές, γιατί μας σώκαρε πολύ. Οι αριθμοί, τα ποσά που θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο των 28 με τιμές 2019 από 2014 με ένα μελλοντικό πλαίσιο με προϋπολογισμό της τάξης του 2%. Θέλουμε πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για το ε, τρέχον πλαίσιο με σταθερές τιμές του 2018 χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε αυτά τα αριθμιστικά στοιχεία και να τα συγκρίνουμε. Γιατί αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία θα μπλέξουμε πάρα πολύ και θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Μερικοί καταφέραμε να τα βρούμε. Ε, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε. Πολλέ ερωτήσει έχω. Χθε τα είπαμε στην Ολομέλεια για κάποια προγράμματα. Λέτε ότι το Erasmus Plus διπλασιάζεται. Θα ήθελα όμω να ρωτήσω. Γιατί έχω καταλάβει ότι υπάρχει και ένα τμήμα του Interrail που συμπεριλαμβάνεται στο Erasmus Plus. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο τμήμα από αυτά τα καινούργια χρήματα θα πάει στο Erasmus Plus και ποιο θα πάει στο Interrail. Δεύτερον, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ποια είναι η πραγματική περικοπή σε σύγκριση με το σημερινό ε, πολιετές πλαίσιο και ιδιαίτερα στο νέο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πόσα κονδύλια θα έχουν τα νέα προγράμματα. Γιατί δεν, αν δεν απατώμε, χάνεται η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και μπαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να χρηματοδοτηθεί. Αλλά υπάρχει και η μέρημνα για τους μετανάστες. Δηλαδή, έχουμε ένα περι κομμένο ε, πώς να το πω, κοινωνικό ταμείο που καλείται να καλύψει περισσότερες αρμοδιότητες. Ε, άλλη ερώτηση. Το νέο ταμείο, InvestEU, αυτό πώς θα λειτουργεί και τι στόχους θα έχει υποτίθεται. Ε, άλλη ερώτηση. Ε, όλες οι διευκολύνσεις και τα καταπιστευματικά ταμεία που είναι εκτός προϋπολογισμού, τι θα γίνουν. Θα χαθούν, θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό. Ποια θα είναι η μοίρα τους. Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο. Ερεσιμότητα. Περισσότερες προφορίες θα ήθελα για το πώς θα λειτουργήσει και αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι οι κυρώσει αυτές δεν θα πλήξουν τους τελικούς δικαιούχου όπως είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Και τελευταία ερώτηση. Περισσότερη ενημέρωση για την ευελιξία. Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστώ. κύριο Μπέντ Κούλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Εννοείται ότι διαφέρουν οι αξιολογήσεις σε διάφορους τομείς. Εγώ αφενός συμφωνώ με την γενικότερη κατεύθυνση, παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για μεγαλύτερη διαφάνεια και όταν έχουμε δύο περισσότερους τίτλους, είναι σημαντικό να καταλαβαίνω πολίτης που πάνε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είναι αυτό πολύ σημαντικότερο στο μέλλον το θέμα της ε, διαφάνειας. Εκεί όπου εξακολουθώ να έχω κάποια προβλήματα είναι με το θέμα πως θα έπρεπε να γίνει ένα πρώτο βήμα όσον αφορά έναν προϋπολογισμό με βάση την απόδοση για συγκεκριμένους τομείς. Να σκεφτούμε τι μπορούμε να θέσουμε ως μετρήσιμους στόχους και να είμαστε αρκετά θαραλέοι να τους καθορίσουμε, να μετράμε και να δούμε. Είμαστε επιτυχείς, πετύχαμε αυτό το οποίο είχαμε καθορίσει ως στόχο ή τουλάχιστον είμαστε στον ε, σωστό δρόμο και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοχή από πλευρά των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν πού πάνε τα λεφτά τους και δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι έχουμε προγράμματα και εντός των προγραμμάτων δίνουμε το 100% των χρημάτων και άρα είναι επιτυχία. Είναι λογιστική επιτυχία και μπορούμε να πούμε ναι εντάξει, αλλά στην ουσία το θέμα είναι τι προκύπτει από αυτά τα μέτρα. Και εγώ εδώ πέρα θα ήθελα να αφαιρθώ στο θέμα της μεταναστευτικής ε, πολιτικής. Εγώ θεωρώ ότι για τη μεταναστευτική πολιτική αφενός ε, χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια αν το δούμε το θέμα ευρύτερα και περιλάβουμε δηλαδή το ότι γίνεται από χώρες ε, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή που χρειάζονται βοήθεια, η οποία κοστίζει. Αλλά ταυτόχρονα, και το λέω, θεωρώ ότι θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να είναι υπό όρους, δηλαδή να υπάρχει μια αποτελεσματική πολιτική ασύλου Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν. Εγώ θεωρώ πράγματι ότι είναι εξαιρετική η αύξηση του προσωπικού της ε, Frontex. Αλλά βεβαίως εξακολουθούν οι άνθρωποι να έχουν το πρόβλημα όταν έρχονται οι πρόσφυγες τι τους κάνουμε όταν δεν έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου του ποιος μπαίνει και ποιος όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς πάμε με βάρκα την ελπίδα και ε, πραγματικά ελπίζω να έχετε την ε, φιλοδοξία αυτή. Αλλά συνολικά νομίζω ότι πηγαίνετε προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το Άλντε η συζητήτρια, κυρία Γιάτεμάκη. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και την ε, σκληρή δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια. Είναι νομίζω δύσκολο να γίνει μία ισορροπημένη πρόταση. Ε, η δική μου ερώτηση αφορά το κλίμα και την ενσωματωσή του της δαπάνες. Εσείς μιλάτε για αύξηση της φιλοδοξίας και να φτάσει το θέμα του κλίματος να είναι 25% των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το τωρινό πι είχαμε έναν στόχο 20% κάτι το οποίο δεν πετύχαμε τελικά. Οπότε, καλοδεχόμενη η πρότασή σας, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εσείς και η Κομισιόν θα πετύχετε τον νέο στόχο, γιατί τον προηγούμενο δεν τον πετύχαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και πάλι σκιώδης από τους Πρασίνους, ο Γιώργη Σολέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, τα καλά νέα από την πρότασή σας είναι ότι δεν είναι οπισθοδρόμηση σε σχέση με το σημερινό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάλι καλά δηλαδή, καλή αρχή είναι αυτή. Τα κακά νέα όμως είναι ότι <laughs> τα χειρότερα θα έρθουν, είναι ακόμα μπροστά μας. Τώρα έχουμε ατέρμονες διαπραγματεύσεις να περιμένουμε, που ελπίζω να μην διαρκέσουν 28 μήνες, όπως την περασμένη φορά. Αλλά μπορεί το τελικό αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων να κάνει κάτι που θα βελτιώσει την πρότασή σας. Εμείς από το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε. Η ομάδα μου θα υπερασπιστεί τη θέση στην οποία καταλήξαμε σε ευρία πλειοψηφία μετά από την έκθεση πρωτοβουλίας. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξη πρέπει να σας πω η πρότασή σας από πλευράς μεγέθους 1,114 δεν νομίζω ότι θα φτάσει για να αναπτύξουμε πραγματικά μια φιλο, φιλόδοξη ε, πολιτική ε, ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα Το ξέρω ότι δεν θέλει μια πολιτικά φιλόδοξη Ευρώπη, ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο, ούτε τμήματα του Κοινοβουλίου. Αλλά είναι μια χαμένη ευκαιρία να δώσουμε περισσότερους πόρους σε μια Ευρώπη καλύτερη, ισχυρότερη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο φιλόδοξη. Η πρότασή σας είναι πιο φιλόδοξη ε, για τα ε, έσοδα και λιγότερο για τις δαπάνες. Βλέπουμε καινοτόμε προτάσεις για τους ιδίους πόρους, για τα έσοδα γενικά, ε, καλοδεχούμενες αυτές οι προτάσεις για τους νέους ιδίους πόρους, αν και θα περιμέναμε ακόμα περισσότερους νέους ιδίους πόρους και άλλου είδους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σωστό βήμα ή ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τις προτεραιότητες, χαίρομαι που εστιάζεται σε πολιτικές στραμμένες στο μέλλον, καινοτομία, έρευνα, ψηφιακή Ευρώπη, Εράσμος, Όλα αυτά είναι πολύ θετικά πιστεύω. Δυστυχώς θεωρείται την άμυνα ως νέα προτεραιότητα όπου θα δαπανίσετε και 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ χρειάζονται χρήματα για την ενεργειακή μετάβαση, για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Νιριάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Χαίρομαι που είπατε ότι επιζητάτε επικριτικά σχόλια. Ελπίζω να δεχτείτε λοιπόν τις κριτικές και στο κενθερμό. Ήθελα εδώ να κάνουμε κάποια αλλαγή και μια διαρκή αλλαγή για το Εράσμος λοιπόν. Είπατε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αρκετή αύξηση, θα θέλαμε ακόμη μεγαλύτερη. Διότι αν θέλουμε να έχουμε κάποια σχέση με την νεολαία μα, να στηρίξουμε τα πανεπιστήμια μα που δεν προχωρούν, του ερευνητέ μα που δεν παίρνουν αρκετά, θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, Ευρώπη που θέλουμε να είναι ευφυή σε μια τέτοια. Χρειάζονται περισσότερε επενδύσει σε αυτή την περιοχή. Επίση, στήριξη χρειάζεται και στον τομέα τη γεωργία για του μικρού γεωργού που έχουν ανάγκε και τι οικογενειακέ επιχειρήσει ε, στη Γεωργία. Εκεί πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερου νέου. Και η περικοπή του 5% στην ε, κοινή γεωργική πολιτική είναι παράδειγμα. Και Πρέπει να κοιτάξουμε να τα ρυθμίσουμε τα ταμεία συνοχής και γεωργίας για να μην ε, παραμείνουν αυτές οι ανισότητες διαρκείας και να υπάρχει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Πρέπει επίσης να πω ότι για, την, ε, για τον κλάδο της αλληλείας αντιμετωπίζει μεγάλες ανάγκες και μεγάλες δυσκολίες ε, μεταξύ των οποίων το Brexit που δεν έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι θα περάσουν ολόκληρη υπεξιακή κρίση. Υπάρχει ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος που χρειάζεται στήριξη λοιπόν. Αν πραγματικά δεν σταθούμε στο πλάι τους με βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο δεν θα πετύχουμε κάτι υγιές για το μέλλον. Εκεί χρειάζονται επενδύσει. Και κάτι άλλο, Επίτροπε, που με απασχολεί πολύ διότι αναγγείλατε την συγχώνευση κάποιων προγραμμάτων. Ξέρουμε ότι αυτό πολλέ φορέ δημιουργεί σχέσει συνεργασία μεν, αλλά πολλέ φορέ και αναπόφευκτε περικοπέ. Και ένα άλλο είναι η χρήση του χρέου ω μόχλευση. Ε, γιατί με την επιφύλαξη τη ε, λιτότητα, και ξέρετε ότι έχουν παραμείνει κάποια στοιχεία αυτή, θα πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι η ειρήνη. Διότι νομίζω ότι οι πόροι για την αμυντική βιομηχανία, την ε, κλείνει και την φύλαξη των συνόρων είναι κάτι, αλλά δεν είναι προτεραιότητα μόνο για το δικό μου κράτο μέλο. Πώ θα πάω, ε, Επίτροπε, στο κράτο μέλο μου και θα πω ε, στου γεωργού, α πούμε, ξέρετε τι αποφάσισε η Ευρώπη. Αποφάσισε να σα αγνοήσει και να δώσουμε λεφτά στη στρατιωτικοποίηση και την άμυνα. Ενώ δεν μα ενδιαφέρει η επιβίωσή σα. Ε, τι θα πούν οι οικογένειε αυτών των γεωργών που είναι αρχοκοκαλιά τη οικονομία μα. Πώ θα απαντήσω στι ερωτήσει του. Πώ θα απαντήσω στου νέου που ε, θέλουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, να να έχουν ε, μια βασική εκπαίδευση. Και εγώ θα τους πω ότι δίνουμε δισεκατομμύρια για την άμυνα, αλλά το μέλλον σας δεν είναι δική μας προτεραιότητα. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση από εσά πώς να το απαντήσουμε αυτό στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας. Ε, διότι αν θέλουμε να ε, συμμετάσχουν στο εγχείρημά μας οι συμπολίτε μας, πρέπει να είμαστε λίγο πιο κοινωνικά, να επιτρέψουμε την κοινωνική συμμετοχή. Και θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμμετείχα στην επεξεργασία πολλών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε μόνο δύο λεπτά, δεν αρκούν. 5% περικοπές για την κοινή γεωργική πολιτική προκαλεί ανησυχίες αυτό. Διάβασα ότι θα υπάρξει μια σταδιακή προσέγγιση βαθμιδών και όχι γραμμική, αλλά παρόλα αυτά οι ανησυχίες παραμένουν και στην συνοχή. Εκεί οπωσδήποτε πρέπει να δούμε να υπάρχει βαθμία προσέγγιση, διότι υπάρχουν οι ε, ε, πιο απομακρυσμένε περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα της και εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε κάλυψη. Είναι ε, σημαντικό για να το καλύψουμε και εντό τη ε, Ευρωζώνης και εκτός και επίσης για την στήριξη της μεταρρυθμίσης. Είναι σημαντικό ε, να δούμε τι μεταρρυθμίσεις θέλουμε να κάνουμε πρώτες, διότι οι μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη μισθολογική υποτίμηση, όπως ζήτησαν τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα προσαρμογής που έχουν εφαρμοστεί, εκεί ε, είμαστε σε τελείω διαφορετικό δρόμο και σε ό,τι αφορά το Ταμείο Σταθερότητα, μάλλον. Ε, και εδώ αυτά τα 30 δι με μια αιρεσιμότητα και έναν πολύ μικρό και περιορισμένο μηχανισμό σταθερότητα. Θέλω να καταλάβω πώ θα ε, χρηματοδοτηθούν όλα αυτά οι κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Τριγκετή Τράπεζα πώς θα πάρουν τα κονδύλια αυτά για να τροφοδοτήσουν του εθνικού προπολογισμού. Δεν θα χρειάζονται εθνικέ προσπάθειε κάποιων κρατών, συγκεκριμένων αυτών τη Ευρωζώνη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε πώς θα συναρθρωθούν αυτές οι προσπάθειες με τις εθνικές, διότι μιλάμε για κάποια δις ευρώ που θα βαρύνουν τα μεγαλύτερα κράτη. Και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, και εδώ σημαντικό πακέτο, 27,5 δις, πρέπει όμως να καταλάβουμε πώς ε, θα διοργανωθούν αυτές οι ομαδικές προμήθειες. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτές θα ωφεληθούν περισσότερο. Εκεί πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποια θα είναι τα κριτήρια απόδοσης ε, για να επιλογούν ε, οι ανάδοχοι από τις διάφορες αμυντικές βιομηχανίες των διαφορών χωρών και για τις ποσοστώσεις ε, εκπομπών άνθρακα. Και εδώ πόροι που θα του ε, διαχειρίζονται οι εθνικοί προπολογισμοί. Αλλά περικοπή του 20% σημαίνει ότι θα πάρουμε κάποια κέρδη από του εθνικού προπολογισμού, κάποια εισοδήματα. Άρα πώ θα το εγκρίνουν αυτό τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση, γιατί με του κανόνε που ισχύουν για τον προπολογισμό είναι δύσκολο να ανακτήσουμε αυτού του πόρου από το εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Βάλη. Ο Αντρέ <clears throat> Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Έτιγκερ. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Φαίνεται πως ε, έχουμε έναν ε, προϋπολογισμό 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, τα σχέδια για Ευρωπαϊκό Στρατό είναι για μας τελείως περιτά, απαράδεκτα και παρεμβαίνουν στην κυριαρχία των κρατών μελών. Ο προπολογισμό αυτό σημαίνει ότι η Ολλανδία θα πρέπει να πληρώνει 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από 7 που πληρώνει αυτή τη στιγμή. Λεφτά τα οποία αφορούν μόνο τι φιλοδοξίε αυτή τη ε, Κομισιόν, οι οποίε δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα. Έχω λοιπόν κάποιε ερωτήσει. Γιατί δεν γίνεται κάποια οικονομία στους μισθούς ε, των υπαλλήλων ε, και των Ευρωβουλευτών γιατί δεν καταργείται η έδρα του Στρασβούργου και αν είστε έτοιμοι να κάνετε οικονομία σε ε, το να σταματήσετε την ε, συνεχώς επεκτηνόμενη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δίνει λεφτά στην Αφρική που δεν πιάνουν κανένα τόπο και στην Ισλαμιστική ε, δικτατορία της ε, Τουρκίας. Θα πρέπει λοιπόν η Ολλανδία να δίνει λιγότερα λεφτά σε αυτό το αποτυχημένο σχέδιο. Το μόνο θετικό είναι ότι έτσι φαίνεται όλο και πιο κοντά τον έξιτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχω τέσσερις ακόμα συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Σιλουάγα. Συγγνώμη, λάθος κάνατε μάλλον. Γιατί η Μαρή Πιέρ είχε ζητήσει πρώτα το λόγο. Μαρή Πιέρ, okay. Ζήτησε το λόγο η Μαρή Πιέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Μαρή Πιέρ Βιού. Ε, βρίσκεται λίγο έτσι εξαπίνης, ε, αλλά ε, θα τα βγάλω πέρα. Ορίστε. Συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρος. Εγώ δίνω το λόγο σε εκείνον που το ζήτησα. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Ναι, μα δεν ζητήσατε να μιλήσετε. Έχει ζητήσει ο κύριος Ιλουάγκα και σας έδωσε εσάς το λόγο χωρίς να το έχετε ζητήσει. Α, το ζητάω τώρα. Παρακαλώ. Ε, ε, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να προσυπογράψω τα όσα υπόθηκαν. Μείον 5% στις άμεσες ενισχύσεις για τη Γεωργία ε, ενώ εντείνονται οι πολιτικές ελευθέρων συναλλαγών. Πώς θέλετε να λύσετε αυτή την εξίσωση με μια γεωργία κοντά στους πολίτες, με εισόδημα δίκαιο και ε, με τρόφιμα ποιοτικά, ε, δηλαδή μικρή γεωργία. Ο συνάδελφός σας Φιλ Χόγκαν δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να καλύψουν τη διαφορά αν θέλουν. Ναι, εντάξει, αν το δούμε έτσι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η κοινωνική πολιτική. Ε, θα μπορούσα ε, αντίστοιχα να σας αποδείξω τι γίνεται με την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Νομίζω ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι η μεταφορά ε, με λογιστικούς όρους μιας πολιτικής σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Συμφωνώ για το Εράσμος αυτά που λέτε, αλλά λιγότερο συμφωνώ με τα όσα είπατε για την άμυνα, την ασφάλεια, τους ελέγχους των συνόρων κλπ. Ερωτώ, Εσεί θέλετε να εξασφαλίσετε, λέτε, το μέλλον της Ευρώπης, αλλά την Ευρώπη για ποιον. Σε κάθε περίπτωση ακούγοντά σα, δεν έχω την εντύπωση ότι θα είναι μια Ευρώπη για όλους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρβαμά. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια έκφραση που σε πολλές γλώσσες χρησιμοποιείται ότι πολύ λόγος γίνεται ε, συνήθως για αυτό το οποίο πιο πολύ λείπει. Μας λείπουν λοιπόν εδώ ακόμα πολλές πληροφορίες όπως είπαν ε, και πολλοί συνάδελφοι. Πάντως να πω τα εξή ότι πρώτον συμφωνώ με τις προτεραιότητες και χαίρομαι για αυτές. Είναι ευρωπαϊκό το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο και με χαρά θα το προσπιστούμε. Αλλά έχω και ένα-δυο ενδιασμού Στο κεφάλαιο 6, γειτονία και ο κόσμος δεν έχει ακόμη τη στρατηγική ε, αξία που του αρμόζει. Αυτό θα το δούμε σε 20 και 30 χρόνια τι μπορεί να σημαίνει. Και δύο, επενδύσεις στις υποδομές. Η ψηφιακή οικονομία είναι άκρο σημαντική, ε, έχει πάρει διαστάσεις όπως και θα έπρεπε, αλλά να μην ξεχνάμε την συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία των διευρωπαϊκών δικτύων Ξέρω ότι θα φτάσουμε και εκεί, αλλά πουθενά δεν το βλέπουμε στην πρόταση πλαίσιο. Το TNT και το SEF, το, ε, τη διευκόλυνση για την Ευρώπη και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ξέρω επίσης ε, και ε, ότι στην πρόταση έχουμε θέλουμε δεσμεύσεις ε, για τους υποχρεώσεις, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιορισμένοι πόροι. Δεν μιλάμε λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Χρειάζονται επενδύσεις και χρειάζεται και χρηστή οικονομική διαχείριση και κατός δικαίου. Μπράβο σας, αλλά εδώ το έχουμε συζητήσει και το έχουμε επιδιώξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι προφανώς ένα από τα σημεία κλειδιά και τέλος, ε, Πρόεδρε, το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα είναι υψής σημασίας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και να φροντίσουμε να γίνει μέσα στη φετινή χρονιά. Ε, μέχρι το τέλος της χρονιάς πρέπει ε, να περάσει το μήνυμα και προς τα κράτη-μέλη μας. Πρέπει να τα πιέσουμε να το καταλάβουν, διότι θα χάσουμε όλοι αν δεν γίνουν όλα αυτά μέσα σε 11 μήνες. Ευχαριστούμε κύριος Μάνκα για ένα λεπτό παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας επενέσω για το ότι χτες και σήμερα είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κοιτάει μόνο τις ε, δαπάνες αλλά και τα έσοδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όσον αφορά τους νέους πόρους. Βρήκα τρεις νέους πόρους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκέφτεστε κι άλλους, γιατί η ομάδα Μόντι περιέλαβε στην έκθεσή της κάτι το πολύ σημαντικό. Για την ε, Συμφωνία των Παρισίων χρειαζόμαστε κάποια μέσα και ένα από τα μέσα στην έκθεση Μόντι ήταν αυτό το οποίο έλεγε ότι θα φορολογούμε τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ε, και οι δασμοί αυτοί θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν αυτό το οποίο προτείνεται εσείς ε, ως ε, ίδιους ε, πόρους και δεν το βλέπω αυτό. Και θα μας βοηθούσε επίσης να προστατεύσουμε και το κλίμα. Επίσης χτες στην Ολομέλεια εγώ αντιληφθήκα ότι οι επενδυτές θα σκέφτονταν μια μεγαλύτερη συνεισφορά στην συνοχή, κατάλαβα καλά. Και μία άλλη ερώτηση. Ο ΦΠΑ θα είναι επιλέξιμη δαπάνη στο μέλλον, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, οι χώρες ε, με έσοδα από ΦΠΑ. Κύριε Σουστοφόρου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όλοι μα και στην Ολομέλεια και εδώ μιλούμε για ισχυρή Ευρώπη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι χωρί ισχυρό προπολογισμό δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη. Και όλοι υπερασπιζόμαστε και υποστηρίζουμε περισσότερα κονδύλια για του νέου, για του αγρότε, για την κοινωνική συνοχή. Πολύ ορθά ο αγαπητό συνάδελφο ο Τζοζέ Μανουέλ Φερνάντε ανέφερε για εδαφική και κοινωνική συνοχή. Αλλά όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε για μικρομεσαίε επιχειρήσει ότι δεν μπορούν να διασφαλιστούν εάν η Ευρώπη δεν έχει αυτοδύναμη άμυνα και ασφάλεια, αν δεν ενισχύσει τα εξωτερικά τη σύνορα, εάν δεν μπορεί η Ευρώπη να διαφυλάξει και να προστατεύσει την κυριαρχία των χωρών μελών πολύ ορθά προχωρούμε σε μια ισχυρή νέα αναμυντική πολιτική και δίνουμε χρήματα για την ασφάλεια. Η ασφάλεια σήμερα αναδεικνύεται ω μείζο ζήτημα. Όμω, όταν μιλούμε για κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ρήτρε των προπολογισμών που αυτόματα θα αποκόπτονται προενταξιακά κονδύλια σε χώρε όπω την Τουρκία, που δεν εφαρμόζει το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει επιτέλου σε αυτά τα ζητήματα να υπάρξει άμεση απάντηση και από εμά εκ μέρου του προπολογισμού, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο Πολλέ φορέ εδώ συζητήσαμε ότι η γραφειοκρατία κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικά δισεκατομμύρια. Ιδού ένα σημαντικό τρόπο μειώνοντα τη γραφειοκρατία να αυξήσουμε τα έσοδα του προπολογισμού. Merci, Monsieur Ευχαριστούμε κύριο Βιώτη πολύ γρήγορα. Δύσκολο να είμαι τόσο γρήγορο, αλλά ευχαριστώ τον Επίτροπο που βρίσκεται εδώ καταρχά. Υπάρχουν θετικέ πτυχέ οι οποίε έχουν ήδη αναπτυχθεί. Θα επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα όμω που για μένα είναι θεμελιώδου σημασία. Πώ σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Ευρώπη στους Ευρωπαίους πολίτες την ιδέα της Ευρώπης που τους φροντίζει με περικοπές στην συνοχή. Περικοπές που σημαίνουν περικοπές και στο κράτος πρόνοιας. Κάτι για το οποίο οι κυβερνήσεις ε, φαίνεται να προσπαθούν να το εφαρμόσουν στην πράξη, το welfare που, όπως λέγεται, το κοινωνικό κράτος. Και μετά για την άμυνα. Εντάξει, αλλά πάρα πολύ ασφάλεια, υπερβολικά πολύ ασφάλεια. Είμαστε υπερ, είμαι υπέρ της άμυνας προσωπικά, αλλά εδώ ε, για τα επόμενα 7 χρόνια να έχουμε τέτοια μεγάλη προτεραιότητα θα έπρεπε να έχουμε προσέγγιση πολύ διαφορετική. Βοήθεια, ναι. Να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης όμως. Όσο για τους ίδιους πόρους δύο ερωτήσεις. Νομίζω δεν ήταν αρκετά τολμηρή η πρότασή σας. Έπρεπε να αυξηθούν σε αριθμό οι ήδη πόροι, όπως είπε και ο συνάδελφος Μάνκα, αλλά να αυξηθούν και σε ποσότητα, σε όγκο. Εκεί πιστεύω ότι μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγο το 12% παραπάνω. Και τελευταίο ερώτημα για τις επιστροφές. Και εδώ υπάρχουν ε, θέματα που θα πρέπει να ξαναδούμε και γρήγορα για τις εκτόσεις. Ευχαριστώ. Αλλά κύριε Τάραντ, σας δίνω μόνο 30 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και την απάντηση. 30 δευτερόλεπτα. Okay. Δεν καταλάβατε. Κύριε Τάραντ. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ που μας ε, παρουσίασε αυτή την υπέροχη πρόταση. Διότι ξέρετε πόσες ερωτήσεις, απαντήσεις και ανησυχίες είχαμε. Τώρα επιτέλους μπορούμε να εργαστούμε. Αλλά τα πάντα, όπως είπε και ο κύριος Σάβαρμα, είναι ε, το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα. Δεν ξέρω εάν ε, στην Επιτροπή είχατε ετοιμάσει ένα πάκο από έγγραφα με όλους τους αριθμούς. Θα είχαμε αρχίσει αμέσως να εργαζόμαστε. Αλλά τέλος πάντων και στις αρχές Ιουνίου καλά είναι να ξεκινήσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση αν θέλετε το θέμα να περάσει από το Κοινοβούλιο και να εγκριθεί φέτος θα πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν είμαστε μονικοί. Θα κάνουμε κάθε τι που περνάει από το χέρι μα για να προλάβουμε μαζί σα και να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μάλετιτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε, Επίτροπε. Ευχαριστώ για το υλικό που έχετε ετοιμάσει. Έχω τρει παρατηρήσει. Η μία έχει να κάνει με τη νέα δομή. Εντάξει, προσπαθήσατε να το κάνετε πιο φιλικό προ το χρήστη και βλεπτό για του πολίτε. Όμως νομίζω ότι και πάλι παραμένει ένα μείγμα ιδεωδών, προγραμμάτων, μέσων, στόχων, αποστολών και δεν είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή είχε μια ξεκάθαρη ε, εικόνα του τι θέλει να κάνει και πώς να φτιάξει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έπειτα, για τα στοιχεία που μας δώσατε αρχικά, αρχικά είναι καλά, λεπτομερή, ωραία τα έχετε πει, αλλά χρειάζεται ο συγκριτικός πίνακας πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το πλαίσιο 2014-2020 για να τα συγκρίνουμε. Και το τρίτο μήνυμα αφορά τις φιλοδοξίες μας. Πραγματικά περίμενα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει με το 1,3 και όχι με το 1,14, διότι το μήνυμά μας το 1,114. Δηλαδή το μήνυμά μας ε, είναι ότι θέλουμε την Ευρώπη σε πρωταγωνιστική θέση στο διεθνές προσκήνιο. Αν θέλαμε να γίνει αυτό έπρεπε περισσότερο να επενδύσουμε στην συνοχή και τη γεωργία και όχι λιγότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, δύο λόγια μόνο για το Εράσμος κύριε Επίτροπε. Το διπλασιάζεται. Σήμερα το Εράσμος είναι μια μηχανή που παράγει βατέωση και ε, το ένα στα δύο αιτήματα απορρίπτεται. Μιλήσατε για, για φοιτητέ. Εμείς θέλουμε και μαθητεία και στην επαγγελματική κατάρτιση και οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι να παίρνουν υποτροφή από το Erasmus ε, Plus. Οπότε χρειάζεται τρίπλασιασμός. Πολλοί μίλησαν για τη δυσκολία συγκρίσιμότητας των στοιχείων. Μπορούμε να προγραμματίσουμε συνεδρίαση των συνεργατών μα, πολιτικέ ομάδε, η Γραμματεία της Επιτροπή, των προπολογισμών, οι δικοί σα συνεργάτε, κύριε Επιτροπή, για να δούμε από την αρχή τη επόμενη εβδομάδα να γίνονται ε, συνεδριάσεις, να τα βάλουν κάτω από τα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πακέτο μας, η δέσμη αυτή, έχει κατατεθεί ε, στα γραφεία σας εδώ και 26 ώρες. Για βγάλτε, 8 ώρες κοιμάστε, μία ώρα τρώτε, μία ώρα ντύνεστε, μία ώρα κάνετε μπάνιο, μπορεί να τα διαβάσετε όλα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε απαντήσει όλες ε, τις ερωτήσεις, θα τα έχετε απαντήσει μόνοι σας άμα τα διαβάσετε. Προφανώς είναι τεχνικές πολλές συνεδριάσεις με ε, τους συνεργάτες, ε, τα γραφεία των βουλευτών, πολιτικές ομάδες, ε, όσες συνεδριάσεις θέλετε, αν θέλετε να τα δούμε ε, άμα θέλετε να έρχομαι όποτε θέλετε. Και τον Αύγουστο. Θέλετε να έρχομαι εδώ τον Αύγουστο, να έρθω τον Αύγουστο. Ε, δεύτερον, ε, σας υπόσχομαι όσο περισσότερη διαφάνεια θέλετε. Και το λέω με κάθε φιλικότητα. Η Επιτροπή γιούνκερ με εμένα επίτροπο θα είναι τόσο ε, διαφανής όπως ήταν η προηγούμενη Επιτροπή Μπαρόζο με Επίτροπο το Λεβαντόφσκι απέναντι στο προηγούμενο Κοινοβούλιο. Δεν κάνουμε τίποτα τεχνάσματα. Μιλάμε για τρέχουσες τιμές και για σταθερές τιμές και τα δύο έχουμε υποβάλει. Έχετε, καν... Έχετε δει την πρότασή μας με δύο καταλόγους πλήρης. Το ένα είναι τρέχουσες τιμές current prices και το άλλο είναι τιμές του 2018. Το ίδιο έχετε και για το σημερινό πλαίσιο, το δημοσιονομικό. Και όλα αυτά μπορούν να αναχθούν σε ένα κονδύλι του προπολογισμού εικονικό με 27 κράτη-μέλη. Δεν ήταν τόσο απλό, καθόλου απλό. Για το Γαλιλαίο ας πούμε. 27 και 28 δεν έχουν διαφορά. Γιατί χρειαζόμαστε τους δορυφόρους και το λογισμικό. Το ίδιο μπορείτε να το υπολογίσετε στη συνοχή και στην κοινή γεωργική πολιτική. Οι Βρετανοί όμως στη γεωργική πολιτική πήραν 15 δισεκατομμύρια περισσότερο από ό,τι στη συνοχή. Δεν είναι λοιπόν η ίδια η στάθμη στη Γεωργία. Μας λείπουν τα 15 δισεκατομμύρια από τη Γεωργία και όχι από τη συνοχή. Όλα αυτά τα λέμε δημόσια. Ποια ήταν η εφητηρία μας ο προϋπολογισμός του 2014-2020, αυτό το PDP. Και το 2020 είναι μέσα, μείον το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό στήσαμε, χτίσαμε έτσι την πρόταση του προϋπολογισμού και κάναμε και τις ε, περικοπές μας, ποσοστία. Περίπου λίγο κάτω από 5% στην κοινή γεωργική πολιτική. Τώρα εξαρτάται από τις ε, εκτελεστικές διατάξεις στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Και τι γίνεται με την εθνική συγχρηματοδότηση στο δεύτερο πυλώνα. Τι γίνεται... Με το τι θα αποφασίσει το κάπινγκ, την οροφή ο κύριος Χόγκαν, την προοδευτική μείωση, για να καταλάβουμε τι θα σημαίνει αυτό για το μικρό αγρότη, για τις άμεσες ενισχύσεις. Ο κύριος Χόγκαν είπε δεν θα πέσει πιο κάτω από 4%. Λιγότερο θα είναι. Θα το δούμε αυτό σε πολλές λεπτομέρειες. Μετά, για τη συνοχή. Τι θα πάρει κάθε κράτος μέλος και κάθε περιφέρεια. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τις εκτελεστικές προτάσεις. Τις εφαρμοστικές. Την περασμένη φορά, στο περασμένο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε μήνες για να τα καταθέσει αυτά. Εμείς είπαμε ε, τέλη Μαΐου θα έχετε τα πρώτα και τα τελευταία 14 Ιουνίου για να γνωρίζουν οι πάντες ποιες θα είναι οι παράμετροι για τη συνοχή. Και τι ρόλο παίζει το ΑΕΠ. Μέχρι τώρα ήταν 86% και τουλάχιστον 80% θα συνεχιστεί στο μέλλον. Ποιο ρόλο παίζει, ξέρω εγώ, η ενεργία, η δημογραφική κατάσταση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή θα σας προτείνουμε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις για να μπορέσετε να αποφασίσετε ποιες παραμέτρους θα επιλέξετε. Αν όμως παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το ΑΕΠ, 86%, θα καταλάβετε ποια επιτυχία θα έχει η συνοχή. Γιατί πολλές χώρες μέλη όταν μπήκαν ήταν κάτω του 60% στο ΑΕΠ του μεσουόρου και τώρα είναι στο 80% και στο 90%. Άρα αυτόματα δεν έχουν αυτές τις ανάγκες που είχαν στο παρελθόν και βγαίνουν. Αυτό είναι επιτυχία της πολιτικής συνοχής, αν έχει φτάσει στο όρο 100%. Θα είναι τα πρώτα νέα κράτη-μέλη που θα φτάσουν στο 100% στην επόμενη προγραμματική περίοδο και μάλιστα το περάσουν κιόλας. Αυτό είναι επιτυχία η περιφέρεια της Βαρσοβίας έχει ξεπεράσει το 100%. Έχει γίνει πια ε, η μηχανή. Ε, δεν είναι η καημένη Πολωνία του 2004. Και σε άλλες περιοχές θα υπάρξουν τέτοιες μετατοπίσεις γιατί επιτυχάνουν τους στόχους και ξεπερνούν το ποσοστό. Αλλά εγώ θέλω κάθε περιφέρεια να ενισχύεται και να υπάρχει και ένα δίκτυο ασφαλείας, ας πούμε. Να μην υπάρχει περιφέρεια που να χάσει πάνω από 30%. Ακόμα και αν υπολογιστικά και λογιστικά λόγω της επιτυχίας της και λόγω ε, της αύξησης του κατακεφαλήν ΑΕΠ ε, θα της αναλογούσε να πέσει στο μείον 40 ή μείον 50%. Σας παρακαλώ κάντε υπομονή λίγες μέρες. Τέλη Μαΐου θα έχετε τα έγγραφα και ελπίζουμε πριν το καλοκαίρι να ξαναβρεθούμε μία, δύο, τρεις φορές όσο θέλετε. Αναφερθήκατε στο θέμα της άμυνας. Να σας πω δύο λόγια στα ράτα γι' αυτό. Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία, Βουλγαρία, όποτε πηγαίνω σε αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα επίσης, ανησυχούν. Ανησυχούν για τη γειτονία. Ο γείτονας εξοπλίζει, εξοπλίζεται. Και η αλληλεγγύη σημαίνει και κοινέ δαπάνες ασφαλείας. Αυτό το σημειώνω. Δεύτερον, το κοινοβούλιο σας, μετά από ε, πρόταση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συμφώνησε και δέχτηκε την Αμυντική Ένωση. Πέσκο, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Τρίτον, πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης είναι και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Και όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν υποχρεωθεί και δεσμευθεί να δίνουν 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Και είναι κάτω του 2%. Και επίσης γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουμε 180 είδη ε, εξοπλισμό, ε, όπλων. Οι Αμερικανοί έχουν καμιά τριανταριά. Και κάθε δολάριο που δαπανούν οι Αμερικανοί πιάνει πολύ περισσότερο τόπο σε λογισμικό, σε όπλα, ε, σε τεθροκισμένα άρματα, πυρομαχικά από ότι οι Ευρωπαίοι, εμείς. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε περισσότερα. 2% κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή για την άμυνα στα κράτη-μέλη είμαστε στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δικό μας πρόγραμμα προβλέπει μέσα σε μια επταετία 13 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια το έτος. Σταγόνες στον ωκεανό σε σχέση με αυτά που δαπανούν τα κράτη-μέλη. Το 1% είναι. Και, ε, μα τι μιλάτε για εξοπλισμούς, αυτά είναι ανοησίες ευρωπαϊκά ε, μέσα θέλουμε, με ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς για να έχουμε οικονομία κλίμακας. Δεν μπορούμε να ε, παραγγελουμε ανταλλακτικά 20 φορές στην Ευρώπη, αλλά μια, δυο, τρεις φορές. Έτσι θα κάνουμε οικονομίες. Έτσι ώστε να μπορεί για το φορολογούμενο να δαπανηθεί και να επενδυθεί κάπου άλλο το χρήμα. Αυτή τη στιγμή είναι αντιοικονομική η κατάσταση στην Ευρώπη που είμαστε τόσο κατακαιρματισμένοι στα αμυντικά. Έχουμε ένα μικρό κεφάλαιο, ένα τίτλο άμυνα και ασφάλεια για να πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματά μας. Και εδώ δεν είναι η άμυνα απέναντι ε, στη γεωργία. Είναι προς το συμφέρον των πολιτών και των φορολογουμένων όλα αυτά. Όσον αφορά τις ε, προτάσεις μας για τους ίδιους πόρους. Είπαμε πως υπάρχει μια θετική διάθεση στο Συμβούλιο για τον ε, ψηφιακό φόρο και θα φέρουμε και τους επόμενους μήνες τους ε, προτάσεις μας. Αλλά να σας υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα τον φόρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τι είχε γίνει. Είχε προταθεί το 2011. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Τι είναι τελικά. Είναι όραμα, είναι μια παρέστηση γιατί όταν ξεκαθαρίσουμε μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για ποιο πράγμα μιλάμε και για ποιες ακριβώς χρηματοπιστωτικές ροές μιλάμε, θα μπορέσουμε να το δούμε και να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές. Θα πρέπει όμως να είναι κάτι το όριμο, όχι σκέψεις οι οποίες δεν έχουν όριμα. Είναι πιθανό να έρθει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο ορισμός του Συμβουλίου. Και θα δούμε το φθινόπωρο, την άνοιξη, τι μορφή θα έχει και θα κάνουμε την πρότασή μας. Θέλουμε το Εράσμος από τα 14 δισεκατομμύρια να διπλασιαστεί και το Interrail μετά από τα 30 εκατομμύρια θα πάει στα 57 α, ε, με στα 30 δις του προγράμματος θα έχει ένα μικρό ποσοστό των 57 εκατομμύριων δεν θα επηρεάσει καθόλου το Εράσμος δηλαδή οι επιστροφές εμείς θεωρούμε ότι μια Ευρώπη χωρίς επιστροφές θα ήταν δίκαιη. Κοιτάξτε δηλαδή, όταν το Λουξεμβούργο έχει η ΑΕΠ κατά κεφαλή 130.000 ευρώ και η Βουλγαρία έχει 6.800 ευρώ ΑΕΠ κατά κεφαλή. Ε, πρέπει νομίζω το 1,1 ως οροφή και στα δύο να είναι ανεκτό. Δηλαδή το Λουξεμβούργο είναι δυνατόν να παίρνει επιστροφή ειδικά αν σκεφτούμε ότι παρόλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό των κονδυλίων επιστρέφει στο ίδιο το Λουξεμβούργο. Η εθνική μα φορολογία είναι προοδευτική όσο περισσότερα κερδίζει κανεί, Όσο περισσότερα έσοδα έχει, τόσο περισσότερο φόρο πληρώνει. Εδώ πέρα, στα δικά μα τα έσοδα τη Ένωση είναι αντιστρόφως προοδευτικό το σύστημα μέσω των επιστροφών. Δεν είναι πάρα πολύ λογικό. Θέλουμε λοιπόν στο τέλο τη περίοδου τα έσοδα μας να προσανατολίζονται στο ΑΕΠ. Και όποιος είναι πιο ισχυρός θα πληρώνει οπωσδήποτε περισσότερο μέσω του 1% ε, αλλά οπωσδήποτε θα ε, κινούμαστε γύρω στο 89-90%. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και αλληλεγγύη με τις ε, επιστροφές. Εδώ πέρα χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου, να εξηγήσω κάτι. Θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει αναστολή πάυση των πληρωμών όπου δεν επηρεάζει άμεσα τον πολίτη. Όταν μιλάμε για εθνικούς εταίρους οι οποίοι είναι παρόλα αυτά υποχρεωμένοι να χρηματοδοτήσουν την πρόταση. Διαβάστε το, διαβάστε το. Είναι πάρα πολύ αναλυτική η πρότασή μας. Και μετά εσείς είστε ο νομοθέτης και μπορείτε να το αλλάξετε. Και αν μου κάνετε κάποια καλύτερη πρόταση θα την δεχτώ. Τώρα εσείς είστε στη θέση του οδηγού. Και έχετε ολόκληρο το πακέτο μπροστά σας. Λοιπόν, τώρα αν έχουμε ιδέες ε, που είναι μακριά από την πραγματικότητα. Εντάξει, σέβομαι την γνώμη σας. Εγώ συναντάω κάθε μέρα κόσμο που έχει τις ανησυχίες και θέλουν να τους βοηθήσει η Ευρώπη εκεί όπου η Ευρώπη είναι η καλύτερη μέθοδος. Μην ξεχνάμε, το, το λιμάνι του Ρότερνταμ ζει από την εσωτερική αγορά. Αν δεν υπήρχαν αγαθά από την κολονία, από τη Βαρσοβία και χωρί εμπορικέ συμφωνίε που έχει συνάψει η Ευρώπη, το λιμάνι της Ευρώπης θα ήταν για ιστιοπλοϊκά, όχι για τάνκερ και κοντέινερ από ολόκληρο τον κόσμο να πηγαίνουν και να έρχονται στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάτε, από την Ευρώπη ζει, όχι από την παραγωγή του Άμστερνταμ, το λιμάνι του Ρότερνταμ. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα, την αμοιβή των βουλευτών, τα αποφασίζετε εσείς, όχι εγώ. Ούτε το... Αυτά είναι υπόθεση δική σα και του Συμβουλίου, σε καμία περίπτωση της Κομισιόν. Για τη μεταρρύθμιση. Εμεί θέλουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συστάσεις αναχώρα που γίνονται εκεί πέρα να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα, αν θέλετε, για τα κονδυλία. Αλλά ποτέ δεν θα δείτε στι συστάσει μας μισθολογικό dumping. Αυτά είναι υπόθεση των εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων μισθολογικό ντάμπινγκ ποτέ δεν πρότεινε στις εκθέσεις της Κομισιόν. Αλλά για την Ιταλία, ε, την οποία αγαπώ. Κοιτάξτε το εξή, στον εθνικό σας υπολογισμό έχετε 1%, 1 για έρευνα και καινοτομία. 1%. Για την Βάδη Βερτεμβέργη είμαστε περήφανοι για το εξή. Είναι 4,9%. Η Ιταλία με αυτήν την βιομηχανία με τις επιχειρήσεις στην Πρέσα, στο Μιλάνο, στο Τωρίνο, στην Πολόνια. Δεν θα έπρεπε να δίνει περισσότερα για έρευνα και ανάπτυξη. Το Μποκόνι χρειάζεται το Πανεπιστήμιο περισσότερα κονδύλια επιγόντως από την Ρώμη. Και τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για το ότι η φία θα μπορούσε να παράγει 2,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο στην Ηλία και παράγει 600.000. Ε, σχετίζεται αυτό με σχέδιο, με κινητήρες, με ποιότητα, με οτιδήποτε. Αλλά μπορούμε νομίζω να το συζητήσουμε αυτό και στον ε, προπολογισμό του 19. Εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, θέλουμε τώρα 26 ώρες μετά την πρόταση να μπούμε στην συζήτηση. Αλλά πιστέψτε με, τον Οκτώβριο θα δημοσιοποιηθούν όλα τα νούμερα. Να συζητήσουμε τα πάντα και δέχομαι όλες τις ερωτήσεις και την κριτική. Είμαστε διατεθειμένοι για στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, κανείς να μην μπορεί να πει ότι υπάρχει κάπου κάτι το μυστικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση, ακροτελευταία, δέχεστε στις διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Αν είχαν βρεθεί κάποιες συμφωνίες, ας πούμε, η Μεγάλη Βρετανία θα έδινε τίποτα όπως κάνει η Νορβηγία και η Ελβετία. Και με βάση αυτή την υπόθεση, πού θα εγγραφεί η Βρετανική συνεισφορά. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο θέμα της Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Και χαιρόμαστε που οι Βρετανοί ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του από την τρέχουσα πραγματική περίοδο μέχρι το 2020 και στη συνέχεια όταν οι δεσμεύσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων γίνουν πληρωμές. Άρα για το σχέδιο προπολογισμού του 19 και το σχέδιο του προπολογισμού του 2020 μπορεί να βασιστούν σε αυτά τα γερά θεμέλια. Δεύτερον, οι Βρετανοί είναι πρόθυμοι ε, να δώσουν τις τρέχουσες δαπάνες όπως είναι οι συντάξεις κτλ. Για το μέλλον εξαρτάται από εκείνους. Horizon, Europe, αν θέλουν να παραμείνουν μπορούν να πληρώνουν όπως η Ελβετία. Και μετά η Οξφόρδη, το Κέμπρις και το Λονδίνο συμμετέχουν όπως η Ζήριχη και η Βασιλεία, τα πανεπιστήμια. Εμείς ήμασταν υπέρ και θα το προτιμούσαμε. Γαλιλαίο, αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πλοήγηση που είναι καλύτερη από την Αμερικανική να μείνουν, αλλά να βάλουν και το χέρι στην τσέπη. Αυτή είναι η συνεργασία για το μέλλον. Τώρα, συνεργασία αστυνομική, μυστικών υπηρεσιών, ε, αμυντική. Ξέρω εγώ, έχουμε πολλές αμοιβαία υποφελεί καταστάσεις όπου και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η Νορβηγία και η Ελβετία θα πληρώνουν στον προπολογισμό, αλλά θα απολαμβάνουν και τις ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες. Άρα, λέει ο Πρόεδρος, θα είχαμε ένα επιπλέον πόρο για τον προπολογισμό, αν ισχύσει κάτι τέτοιο αλλά δεν φαίνονται στον προπολογισμό ε, οι πόροι από την Ορβηγία και από την Ελβετία πηγαίνουν στο Ταμείο Συνοχής. Έχουμε ένα ψήφισμα για το Μάιο το οποίο θα φασιστεί σε αριθμούς όσο γίνεται πιο σαφής. Ερωτώ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τη Δευτέρα να αρχίσουν να συναντιούνται οι συνεργάτες μας για να βάλουν κάτω όλα τα στοιχεία κτλ. Βεβαίως είπα, ναι. Ωραία. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Λήξη συνεδρίασης. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε ραντεβού πολλά θα έχουμε στο μέλλον και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την προθεσμία που δηλώνεται.